αντιρρήσει. Μάλιστα, έτσι επικυρώνονται οι εντολές αυτός. Από τους μη εγγεγραμμένους έλαβα αιτήματα ορισμού στις ε, επιτροπές και στις ε, κοινοβουλευτικές ε, αποστολές. Ο κατάλογος αυτός θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούμε ότι ισχύουν αυτά τα αιτήματα. Θα ήθελα να